Ευρωπαίοι χαίρομαι ιδιαίτερως για την συμφωνία που εξευρέθη. Οι όταν έχουν άδεια μητρότητα, θα χρειάζονται ενδεχομένω ευέλικτη ε, σχέση εργασία. Εάν του προσφέρουμε αυτή τη δυνατότητα θα μπορούν να τα γυρίσουν ταχύτερα στην ε, εργασία τους και έτσι να αναπτύξουν και τις σχέσεις ε, συνδυασμού του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο που είναι απαραίτητε. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να του προσφέρουμε, είναι κάτι από το οποίο στη τελευταία ανάλυση εξαρτώνται τομεί ολόκληρη οικονομική δραστηριότητα. Αν μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερη ασφάλεια, για να μπορέσουμε να δώσουμε ασφάλεια απασχόληση στου εργαζομένου, δεν πρέπει να μειώσουμε την ευελιξία στον χώρο εργασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καλωσορίζω τη βελτίωση που επετεύχθη με, με την εξασφάλιση των ελάχιστων ε, προϋποθέσεων ασφαλείας των ε, εργαζομένων, εκατομμυρίων εργαζομένων στην Ευρώπη που μπορούν να επικαλυστούν μια συνθήκη, μια σύμβαση εργασίας, αλλά δεν καλύπτονται επαρκώς όλοι οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη. Οι επισφαλείς ε, θέσεις εργασίας πρέπει να εξασφαλίζουν περισσότερα δικαιώματα βεβαίω, Μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν από την προσφορά της εργασίας πρέπει να υπάρχει ενημέρωση αλλά, ε, για την ε, καταγγελία, αλλά χωρίς όρια χρονικά. Ε, ένα ζήτημα το οποίο συζητείται πισταμένος στη Γερμανία. Δεν μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε σε σχέση με το Συμβούλιο επαρκής επιτυχίες προστασίας των εργαζομένων και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε είναι ότι εκείνοι οι οποίοι εργάζονται λιγότερο από 32, λιγότερες από 32 ώρες τον ε, μήνα είναι αυτοί οι οποίοι είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στην αυθαιρεσία. Πρέπει η Ευρώπη να κάνει ακόμα περισσότερο για τους εργαζομένους. Ήσασταν κάπως γρήγορος κύριε Ντετιέν. Φιέλνερ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι λίγο σουρεαλιστικό να βρισκόμαστε εδώ όχι για την τελευταία ολομέλεια, γιατί επίσης οι σοσιαλδημοκράτες, ε, ε, οι Σουηδοί λένε, δεν συμβαίνει αυτή η συζήτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ρυθμίζει τη Σουηδική αγορά εργασία και αν το κάνει δεν έχει αυτό σχέση με τον κοινωνικό πυλώνα. Στέφαν Λαβίν, ε, ο Πρωθυπουργό, είπε πως πρόκειται για μύθο. Αλλά αν θέλετε να δείτε τι ακριβώς λέει αυτό το έγγραφο, θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα της Κομισιόν που απορρέει από την διάσκεψη κορυφής του, του το 2017. Αλλά αυτό ε, ε, δεν συμβαίνει. Κάποιες φορές οι σοσιαλδημοκράτες οι Σουηδοί ξυπνάνε όπως πέρσι τον Νοέμβριο που ε, αποκάλεσαν αυτή την πρόταση απαράδεκτη, που σοβαρά θα επηρεάσει το σουηδικό μοντέλο, το σουηδικό πρότυπο με τις συλλογικέ μας συμφωνίες. Είναι σωστό πως ε, ε, συμβαίνει αυτό και είναι απίστευτο που το υπερψηφίζουν. Και πάλι λένε ότι όχι δεν συμβαίνει. Αυτό ίσως και γι' αυτό να λείπουν και δεν, να μην συμμετέχουν, γιατί αυτό που συμβαίνει εδώ φαίνεται να μην συμβαίνει, τουλάχιστον σύμφωνα με τους σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ. Μπαίνουμε στο Κάτσι με την κυρία Γεσλοβιέσκα για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, ε, ζούμε σε καιρούς όπου η αγορά εργασίας αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Α, ξεπηδούν νέα επαγγέλματα και νέες μορφές απασχόλησης. Η ευελιξία είναι σημαντική και για τις δύο πλευρές. Ευέλικτες μορφές απασχόλησης ε, διευκολύνουν την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και οικογενειακής ζωής και για τις επιχειρήσεις πρέπει αυτές να αντιμετωπίσουν την αγορά όπως αυτή αλλάζει. Όμως θα πρέπει να υπάρχουν κάποια μήνυμα μίνιμουμ καθολικά δικαιώματα για τους εργαζόμενους. Έχουμε εργαστεί σκληρά στην Επιτροπή της Απασχόλησης και έχουμε τη λύση. Αυξάνουμε το επίπεδο ασφάλειας. Λίγο πιο αργά παρακαλεί η Πρόεδρος ε, την ομιλήτρια. Μάλιστα. Χωρίς όμως ε, λοιπόν να επιβαρύνονται ε, υπερβολικά οι εταιρείε. Και αυτό γιατί υπάρχουν ιδιαιτερότητες στα κρατημέλη. Εδώ στην οδηγία έχουμε κοινέ απαιτήσει για γραπτές δηλώσεις, για την παροχή ενημέρωσης, γραπτής ενημέρωσης ε, εντός 7 ημερών στη βασική τους μορφή και εντός 30 ημερών με όλες τις λεπτομέρειες. 6-7 μήνες είναι δοκιμαστική περίοδος και αυτό, όπως είπαμε, βελτιώνει πολύ την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ και εγώ σας ευχαριστώ. Curtin Darling. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2016 η Επιτροπή Αναφορών του Σώματος άκουσε τους εργαζόμενους στο McDonald's σε διάφορα μέρη της Ευρώπης για το πόσο επισφαλής ήταν η κατάστασή τους από πλευρά συμβολέου και συνθήκων. Ήταν η εκστρατεία που έκαναν για το unhappy meal Εργάστηκα μαζί τους και με ενέπνευσε αυτά που είπαν οι κυρίως νέοι εργαζόμενοι στην εργασία που εργάζονται στον τομέα αυτό των fast food για να πούμε όχι, αρκεί, θέλουμε αξιοπρεπή συνθήκε εργασία και αξιοπρεπή αμοιβή. Και κάνουμε ένα βήμα λοιπόν αυτή τη βδομάδα με αυτή την κατεύθυνση. Οι κανόνε για την τις ε, διαφανείς και προβλέψεις συνθήκες εργασίας δεν ε, πηγαίνουν όσο μακριά θα ήθελα. Θα ήθελα να απαγορεύεται συγκεκριμένα το συμβόλαιο το τόσο εκμεταλλευτικό των μηδέν ωρών και να υπάρχει εκπεφρασμένα κάλυψη όλων των εργαζομένων ανεξάρτητα από το αν είναι δημόσιοι πάλι ιδιωτικοί και ανεξάρτητα από τον αριθμό των ωρών. Αλλά όπω είπε και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, οι κανόνε αυτοί δίνουν νέα σημαντικά δικαιώματα στου επισφαλεί εργαζόμενου και στου εργαζόμενου με βάρδιε παντού στην Ευρώπη. Οι κανόνε αυτοί πρέπει να εφαρμοστούν πλήρω, χωρί παραθυράκια και εξαιρέσει. Είναι ελάχιστα δικαιώματα. Α κάνουμε περισσότερα. Η αύξηση της επισφάλειας στην εργασία δημιουργεί περισσότερη οικονομική ανασφάλεια, την οποία εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά. Σταματήσουμε αυτή την εκμετάλλευση. Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να εκπροσωπεί την προσπάθεια καλές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κοινωνία μας πρέπει να παρέχει σε όλους τους εργαζόμενους αυτές τις ε, συνθήκες. Πρέπει οπωσδήποτε να, να αντιμετωπίσουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Οι νέοι πιο ευέλικτοι τύποι εργασίας μπορεί να δημιουργήσουν και ευκαιρίες για την ε, ψηφιακή οικονομία, αλλά πρέπει οι εργαζόμενοι να εργάζονται με αξιοπρεπείς συνθήκες. Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουν σωστά δικαιώματα σε μια αγορά εργασίας που είναι σε συνεχή ροή. Πρέπει να υπάρξουν εγγυήσει για τις επιχειρήσεις, να υπάρχει σωστή ισορροπία λοιπόν στη σχέση μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων. Η κυρία Κούνεβα. Πώς θα γίνει να έχουμε διασφαλής και προβλέψιμο όρο εργασία στην ευρωπαϊκή ένωση όταν στερούμε από την πληροφόρηση εκατομμύρια εργαζομένων. αυτό θα κάνουμε αν υπερψηφίσουμε το αποτέλεσμα του τριλόγου θα νομιμοποιήσουμε την επισφαλή εργασία διότι το κείμενο με τις προτάσεις του συμβουλίου δεν ενισχύει την προστασία των εργαζομένων αλλά μόνο την ευελιξία γιατί στηρεί την ενημέρωση που πρέπει να έχουν για τις συνθήκες και το μισθό εργασίας τους από την πρώτη μέρα της πρόσληψής τους. αγνοεί παντελώς ότι πολλοί αυτοαπασχολούμενοι στην πραγματικότητα είναι μισθωτοί. το συμβούλιο δεν έχει καταλάβει τίποτε από την εξέγερση των κίτρινων γυλαίκων στην γαλλία δεν έχει καταλάβει τίποτε από τη φωνή των πρεκαριάτων που σιγά σιγά δυναμώνει σε όλη την ευρώπη. εμείς εδώ οφείλουμε να τους ακούσουμε. ευχαριστώ. Ζητήσατε το λόγο κύριε μου στα πλαίσια του Catch Πολύ καλά. Παρακαλώ λοιπόν, Εσύ τότε. Οι συνθήκε εργασία είναι πολύ σημαντικέ. Γιατί οι συνθήκε εργασία είναι από τα σημαντικά στοιχεία τη ζωή μα. Ω ε, εισηγητή του ΕΛΚ στην Νομική Επιτροπή, εργάστηκα για αυτήν την οδηγία και συναντήθηκα με ενό εργαζομένων και εργοδοτών στην ε, Μάλτα. Και ακούει κανείς απίστευτα πράγματα. Εργαζόμενοι που εργάζονται χωρίς συμβόλαιο. Που δεν ξέρουν πότε θα πληρωθούν για πρώτη φορά. Και επίσης εργαζόμενοι που πρέπει να πληρώσουν για την ε, κατάρτισή τους για να μπορέσουν να εργαστούν. Αυτό ισχύει ακόμη και για δημόσιους υπαλλήλους. Στέλνει λοιπόν ένα σαφές μήνυμα αυτή η οδηγία. Θα πρέπει να βοηθάει όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τις επιχειρήσεις. Γιατί όσο καλύτερες είναι οι ελάχιστε ηθίκε ε, για τους εργαζόμενους, υπάρχει και πιο υγιής ανταγωνισμό μεταξύ όλων των επιχειρήσεων. Η κυρία Ward. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Οι ε, ανθρακορίχοι που ε, έσπαγαν τις μέσες τους ε, δεν είχαν καμία ασφάλεια ούτε και οι εργαζόμενοι στα λιμάνια στο Λίβερπουλ το 19ο αιώνα είχαν καμία προστασία. Πώς όμως τον 21ο αιώνα όπου μπορούμε να πιάσουμε το φεγγάρι, να στείλουμε τον άνθρωπο στον Άρη, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Μέσω της οικονομίας ε, που αλλάζει, της αγοράς εργασίας που αλλάζει μέσω της τέταρτης ε, ε, βιομηχανικής επανάστασης, θα πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους σε αυτό το νέο οικοσύστημα του χώρου εργασίας. Με την Βρετανική κυβέρνηση που ακόμα προσπαθεί να φύγει από την Ένωση και με τον κίνδυνο οι συντηρητικοί να προσπαθήσουν να νερώσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πω η νομοθεσία για προβλέψιμε και διαφανεί συνθήκε εργασία μαζί με τι συλλογικέ διαπραγματεύσει για όλου του εργαζόμενου σε όλα τα 28 κράτη-μέλη είναι ο καλύτερο τρόπο για το Ενωμένο Βασίλειο, για του 27, για τα συνδικάτα και για τι εργατικέ δυνάμει. Ο κύριο Μαριά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε ξανά στο ίδιο έργο θεατές διότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι τελικά επιβεβαιώνει την πολιτική της η ευρωπαϊκή ένωση δηλαδή πρακτικά αφήνει τις ε, εργασιακές σχέσεις στο πεδίο της ευελιξίας στις άτυπες μορφές και επί της ουσίας δεν διασφαλίζει και την μόνιμη απασχόληση και κυρίως ρυθμίσεις οι οποίες πραγματικά να στηρίζουν την ίδια την απασχόληση των εργαζομένων και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα το οποίο έχει η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία που συζητούμε. θέλω να επισημάνω επίσης ότι πρέπει να σταματήσει η υπερεκμετάλλευση που γίνεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους αναπληρωτές δασκάλους και τους αναπληρωτές καθηγητές. χιλιάδες εκπαιδευτικοί είναι σε ομοιρία αυτή τη στιγμή στην ελλάδα δεν ρυθμίζονται οι σχέσεις τους με βάση την οδηγία 1999 δηλαδή να έχουν πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα και να διοριστούν. Είναι ένα σοβαρό θέμα, το συζητήσαμε στην Επιτροπή Αναφορών και πρέπει να ρυθμιστεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι νέες μορφές απασχόλησης, όπως η απασχόληση on demand, απαιτούν μεγάλη ευελιξία ε, και διαθεσιμότητα. Όμως αυτά δεν μπορούν να είναι νέες μορφές ε, φθηνής και επισφαλούς εργασίας που θρέφεται από τους ανθρώπους που μένουν έξω από το σύστημα. Αυτή η οδηγία θα μπορούσε να ήταν πιο φιλόδοξη και για όλους, γιατί ο στόχος της ήταν να δώσει βεβαιότητα στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, αφήνοντας απ' έξω τις μηδενικές συμβάσεις ή αποκλείοντάς τις από τα κεφάλαια ε, των ελάχιστων απαιτήσεων υπηρεσίες επίγουσες εργαζόμενους στην θάλασσα κτλ. Δεν προστατεύει αυτούς που το χρειάζεται περισσότερο και μάλιστα τις γυναίκες, όπως είναι ε, οι οικιακές βοηθοί που κάνουν ένα σωρό εργασίες και προσφέρουν φροντίδα και που μένουν εκτός αυτής της νομοθεσίας. Λίγο πιο αργά παρακαλεί η Πρόεδρος. Έλεγα για τις οικιακές βοηθούς ότι μείναν έξω από, αυτές τις, ε, αυτά τα νομοθετήματα ενώ θα έπρεπε να έχουν περισσότερη αξιοπρέπεια στι συνθήκε εργασία του. Δεν μπορούμε να στηρίξουμε αυτή την νομοθεσία που άδικα αφήνει απ' έξω αυτούς που το χρειάζονται, τη χρειάζονται περισσότερο. Κλείσαμε το καρδιά. η κυρία Τάισεν. Okay. Thank you, Madam President. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, έχω ήδη ευχαριστήσει τον εισηγητή, αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές και τη Ρουμανική Προεδρία για την, τις επιτυχίες διαπραγματεύσεις. Ε, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, η προτινόμενη οδηγία για τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας εστιάζουν σε αυτό που είναι πραγματικά απαραίτητο για τους εργαζόμενους στην σημερινή αγορά εργασίας. Η ευελιξία είναι απαραίτητη όπως και η ψηφιοποίηση και γι' αυτό δεν, προστατε... δεν με να απαγορέψουμε νέου είδους απασχόληση, αλλά να μιλήσουμε για προστασία ενάντια σε υπερβολικές ε, ε, καταχρήσεις, ε, όμως προβλέποντας και ότι όλοι πρέπει να οργανώσουν κάπως τη ζωή τους. Η, η οδηγία αυτή θεωρεί κοινό καθήκον για όλους ότι πρέπει να αφήσουν όλοι αρκετό να, να επιμείνουν ώστε, επί τόπου ώστε να είναι επιτυχή. Θα πρέπει να στηριχθούν τα μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύη για όλους τους συμπολίτε μας. Όπω είπα και παλιότερα, Πρόεδρε, αυτή η οδηγία επίσης είναι μέγα επίτευγμα ώστε η Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων να καταστεί πραγματικότητα. Όλοι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό το ορόσημο. Ε, ξέρετε, κύριε Ευρωβουλευτέ, θέλω να τελειώσω συνδέοντα αυτή την οδηγία και άλλε μα πρωτοβουλίε η απόσπαση εργαζομένων, η προστασία αυτών, η πρόσβαση στην κοινωνική πρόνοιαση για όλους, περισσότερο ευρωπαϊκό εξάμενο και να μην ξεχνάμε και την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Όλες αυτές οι προσπάθειες δείχνουν πως αυτή η Επιτροπή μαζί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουμε καταφέρει πολλά και έχουμε φέρει πίσω την, την κοινωνική Ευρώπη στο επίκεντρο της δράσης της Ένωσης. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Καλβέτ Τζαμπόν για να κλείσουμε το θέμα. Εκ νέου να ευχαριστήσω πολύ, ε, Πρόεδρε. Σέβομαι απόλυτα και είναι οι μόνοι άνθρωποι στους οποίους θα απαντήσω αυτοί οι οποίοι ε, δείχνουν ε, επιφυλάξεις ε, αν τους παρηγορεί αυτό, πράγμα το οποίο δεν το πιστεύω, ε, θα πω ότι και εγώ είμαι μεταξύ αυτών που θεωρούν πως δεν προχωρήσαμε αρκετά, δυστυχώς. Αλλά ε, εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να βρούμε μια ισορροπία. Ε, αυτό που διαπιστώνουμε βασικά είναι τρία σελήψεις. Το πρώτο είναι ότι δεν καλύπτονται όλοι, γιατί ε, απαιτούνται 3 ώρε ε, εβδομαδιαίω και 12 μηνιαίω. Είναι αλήθεια, θα το είχαμε προτιμήσει να καλύπτονται όλοι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πρόοδο σε σχέση με το τι είχαμε πριν. Ε, και εν πάση περιπτώσει να σα θυμίζω ότι ζητήσαμε από την Κομισιόν να επαγρυπνεί ενεργά, ώστε εάν ε, πολλαπλασιαστούν οι συμβάσει των 12 ωρών μηνιαίω, τότε θα πρέπει να λάβουμε μέτρα. Κατά δεύτερο λόγο, επίσης, έχουμε το θέμα των εξαιρέσεων. Δεν τις εγκρίνω, δεν, τις, δεν καταλαβαίνω αυτά τα λόμπια. Ας πούμε, οι εργαζόμενοι στη θάλασσα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπο να βρούμε μια ισορροπημένη συμφωνία χωρίς να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Το λέω με για τη συνείδηση. Και ναι, οι μηδενικέ ώρε. Οι μηδενικέ ώρε μα δυσκόλεψαν πάρα πολύ και είναι μάλιστα από εδώ και στο εξή δεν μπορούν να ανανεωθούν. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν στους συναδέλφους είναι ότι έθεσαν τα θέματα αυτά να σε σκεφτούν. Είναι καλό, ακόμα και αν δεν είναι τέλειο, για, καλό είναι να υπάρχει για το μέλλον για τους Ευρωπαίους εργαζόμενους. Είναι καλύτερο από το τίποτα. Εγώ εκεί κατέληξα και σέβομαι τις φιλοδοξίες και σέβομαι τους ε, ότι καλοπροαίρετα επικρίνουν τον κόσμο. Πάντω πιστεύω ότι είναι καλύτερο από το τίποτα και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μεγάλη στήριξη από ολόκληρο το Κοινοβούλιο σε αυτό το στάδιο τη οικοδόμηση τη κοινωνική πολιτική τη Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ όλους, λέει η Πρόεδρος. Κλείνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα. Περνάμε τώρα στην έκθεση του κυρίου Λέναρς για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας με εσάς κύριε Λέναρς καταρχήν για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά στηρίζεται στην ελευθερική κυκλοφορία των πολιτών, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών απαρτίζουν την ε, εσωτερική αγορά και εξασφαλίζουν την ε, ευημερία για τους πολίτες. Δεν είναι όμως μόνο ελεύθερο εμπόριο και οικονομία Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εσωτερική αγορά πρέπει να είναι μια αγορά δίκαιη. Μια αγορά όπου ο εργαζόμενος θα κερδίζει αυτά που αξίζει, όπου δεν θα πέφτει θύμα εκμετάλλευσης. Δεν πρέπει λοιπόν να υπάρχει εκμετάλλευση, δεν, δεν πρέπει να υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Πρέπει να είναι σε θέση οι επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται πέραν των ε, συνόρων με διαφύλαξη όμως των συνθήκων θεμητού ανταγωνισμού. Μια αγορά όχι μόνο ελεύθερη αλλά και δίκαιη είναι ο όρος που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε. Συνθήκες ισότιμης απασχόλησης, διακίνησης εργαζομένων ε, πολιτών, ε, εμπορευμάτων και πρέπει να εξασφαλιστεί ένας μηχανισμός σεβασμού, επιβολής της ε, τήρησης της νομοθεσίας. Μας έχει απασχολήσει πολύ το θέμα αυτό. Η οδηγία για την απόσπαση, παραδείγματι, που προβλέπει την ε, ίση αμοιβή για, την, ε, για, ίση, για ίδια εργασία, αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο προστασίας των εργαζομένων. Έχουμε προστατέψει τους εργαζομένους σε σχέση με την απασχόληση κατά την οποία χειρίζονται επικίνδυνες ουσίες. Έχουμε κάνει πολλά βήματα για την προαγωγή μιας ε, δίκαιης αγοράρης εργασίας, μιας ισότιμης πρόσβασης στην εργασία. Αλλά αυτό που έχουμε γράψει επί χάρτου δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει στην πράξη να υλοποιήσουμε αυτά που έχουμε προβλέψει. Είναι ε, πολλά εκατομμύρια οι πολίτες οι οποίοι ζουν σε διαφορετικές χώρες από τη χώρα προέλευσης και εργάζονται εκεί και αυξήθηκαν μάλιστα στα τελευταία δεκαετία σημαντικά οι αριθμοί αυτών. Ωστόσο βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς επιθεωρήσεις ε, και έλεγχοι των συνθήκων υπό τις οποίες εργάζονται, κυρίως οι διασυνοριακοί. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν διασυνοριακοί έλεγχοι από τις επιθεωρήσεις εργασίας Σήμερα μπορούμε να δείξουμε πως είμαστε σε θέση να ε, αναλάβουμε την πρόκληση και να φέρουμε αποτελέσματα, αποτελέσματα ικανοποιητικά γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν έχει περάσει ένας χρόνος από την κατάθεση της πρότασης της Επιτροπής αυτό που έχουμε μπροστά μας λοιπόν μας επιτρέπει να εισαγάγουμε νέες συνθήκες εργασίας, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους και κοινέ επιθεωρήσεις ή αυτοψίες ε, αλλά και διαμεσολάβηση μεταξύ των κρατών μελών σε περίπτωση ε, μη τήρησης κανόνων. Μπορούμε να εντοπίσουμε αδυναμίες στα συστήματα για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Όλα αυτά θα τα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, για την προστασία των εργαζομένων μια γνήσια υπηρεσία που μπορεί να καταπολεμήσει με το έργο της και τις ε, ενδεχόμενες απάτες για την προαγωγή της εσωτερικής αγοράς στον χώρο της απασχόλησης και κλείνοντας θα θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Τίσεν για την πολύ σημαντική πρωτοβουλία η οποία κατέστησε δυνατά τα αποτελέσματα για τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Ευχαριστώ δε και την Προεδρία της Ρουμανίας η οποία προέβλεψε με την προσήλωση που τη χαρακτηρίζει ένα πυκνό χρονοδιάγραμμα, ένα σφιχτό χρονοδιάγραμμα για τις συνομιλίες και επίσης μας επέτρεψε να προχωρήσουμε για τους συναδέλφους ε, με τους οποίους συνεργάστηκα τους, ε, τους και πρέπει να σας πω αλλά μην το πείτε στη γυναίκα μου ότι εσάς σας έχω δει πιο συχνά από ό,τι έβλεπα τη σύζυγό μου το τελευταίο διάστημα μην τη το πείτε μόνο ε, ευχαριστώ λοιπόν θερμά για την ε, πολύ καλή συνεργασία και κυρία Πρόεδρε κλείνοντα, ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μας και όλους τους ε, Σύμβουλους που έχουμε στην υπηρεσία μας, χωρίς τους οποίους θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τέισεν για τρία λεπτά. Χαίρομαι πολύ και εγώ που βρίσκομαι ενώπιον σα πριν την ψηφοφορία για τον κανονισμό που ιδρύει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία. Πάντα θεωρούσα ότι αυτό είναι το αποκορύφωμα της νομοθεσίας. Το Μάρτιο του 2018 κατέθεσα την πρόταση και ένα χρόνο αργότερα ήρθαμε να ψηφίσουμε τον τελικό κανονισμό. Είναι εντυπωσιακό αυτό το αποτέλεσμα στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και αυτό δείχνει πόσο σοβαρά παίρνουν την υπόθεση οι δύο συνομοθέτε και πόσο σκληρά εργάστηκαν ο εισηγητή, οι συνεισηγητέ και οι διαδοχικέ ε, προεδρίε του Συμβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή Γιώργον Λέναρτ για την εξαιρετική του ε, προσήλωση όσο και διεύθυνση των διαπραγματεύσεων από πλευρά Κοινοβουλίου. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω του και και την Προεδρία του Συμβουλίου για την επικοδομητική του στάση, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ε, γρήγορα αυτή η υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ε, θα είναι ε, ο πρώτος επιχειρησιακός λειτουργικός οργανισμός στην αγορά εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται οπωσδήποτε να θεσπιστεί σήμερα 17 εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών ζουν ή εργάζονται σε άλλη χώρα από την πατρίδα τους. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Αρχή Εργασίας ε, θα συσταθεί για τους πολίτες αυτούς έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η νομοθεσία και οι κανόνες να εφαρμόζονται με τρόπο ε, συστηματικό, σοβαρό και συνεπή. Είναι τρεις οι στόχοι ίση σημασία. Πρώτον, διευκόλυνση στην πρόσβαση πληροφοριών ε, για επιχειρήσει και πολίτε οι οποίοι όταν ε, μετακομίζουν στο εξωτερικό θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Ο οργανισμός αυτός θα φροντίζει ε, όλοι να τηρούν και να συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς για την απόσπαση εργαζομένων και για την καθημερινή ε, λειτουργία της δικτυακής πύλης Γιούρες, για την κινητικότητα των εργαζομένων. Δεύτερον, η αρχή αυτή θα εξασφαλίσει το συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με την ε, επιβολή του Ευρωπαϊκού Νόμου την κοινωνική ασφάλεια, το συντονισμό της και την κινητικότητα των εργαζομένων. Έτσι θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη στη διασυνοριακή του συνεργασία ε, για την ανείχνευση και την καταπολέμηση ε, των ατασταλιών και της παράνομης εργασίας. Βασιζόμενοι στα παραδείγματα της Eurojust και της Europol, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα συνενώνει εθνικούς εμπειρογνώμονες για την ανταλλαγή ε, πληροφοριών και τη συνεργασία και τη διευκόλυνση όλων αυτών. χωρί καμιά αμφιβολία όλα αυτά θα συνεισφέρουν σημαντικά στη δημιουργία μια ε, κοινή κουλτούρα επιβολή του νόμου με επίσημε ανταλλαγέ εμπειρογνωμόνων και αμοιβή εμπιστοσύνη. Επίση, θα υποστηρίζει και τι εθνικέ αρχέ επιθεώρηση εργασία ε, για ε, συντονισμό, συνεννόηση και κοινέ επιθεωρήσει. Και τρίτον, θα είναι ένα φόρουμ διαμεσολάβηση μεταξύ των διαφόρων αρχών σε περίπτωση διαφορών για εξοδικαστικούς διακανονισμούς έτσι ώστε να δίνονται ταχείες απαντήσεις σε διενέξεις που αφορούν με μεμονωμένους πολίτες ή εταιρείε. Γνωρίζω ότι πριν από μία διετία όταν αρχίσαμε να συζητούμε καν την πιθανή δημιουργία αυτού του οργανισμού ορισμένοι αμφέβαλαν ε, ως προς την προστιθέμενη αξία άλλου ε, ενός ευρωπαϊκού οργανισμού. οι επιχειρησιακές ε, όμως αρμοδιότητες δεν υπήρχαν ακόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τώρα αυτό έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας για την καθημερινή επιβολή των διατάξεων και των νόμων και ταυτόχρονα θα ανοίξει και ευκαιρίες για μια δίκαιη κινητικότητα των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή εγκριθεί η δική μας Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να κάνει τα πρώτα πρακτικά βήματα έτσι ώστε να καταστεί ε, λειτουργικός οργανισμός αυτό μέχρι το φθινόπωρο του 2019. Πραγματικά προσβλέπω και περιμένω να ακούσω τις ε, παρατηρήσεις σας ε, στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Ο κύριος Γκάιερ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη Επίτροπε Τάισεν κυρίε και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία θα ασχοληθεί με την αποτελεσματική και ουσιαστική ε, εφαρμογή τη νομοθεσία στην ευρωπαϊκή κινητικότητα των εργαζομένων. Καλό είναι αυτό. Και θα είναι ο πρώτο συνομιλητή για τι εθνικέ επιθεωρήσει εργασία ε, που καλούνται να κάνουν διασυνοριακού ελέγχου έτσι ώστε να καταπολεμηθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και το μισθολογικό ντάμπινγκ. Πολύ καλό είναι. Και έτσι προστατεύονται και οι νομοταγεί εταιρείε από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Όλα αυτά είναι ωραία. Αυτό που δεν είναι ωραίο είναι ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί πλήρω αυτό ο οργανισμό, παρόλο που είναι σημαντικό ορόσημο. Εμεί θα θέλαμε να έχει περισσότερε ελεγκτικέ αρχέ, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασία, ελεγκτικέ αρμοδιότητε δηλαδή, ε, για κράτη-μέλη που είναι απρόθυμα να συνεργαστούν. Και επίσης δεν συμμετέχουν επαρκώ οι κοινωνικοί εταίροι στη διαχείριση τη εταιρεία. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι φιλελεύθεροι και η συντηρητική ομάδα έχουν ε, προβεί σε αυτή την αμέλεια. Και ελπίζουμε στη διένεξη για την έδρα ε, να πριτανεύσει περισσότερη λογική από ό,τι μέχρι σήμερα. Τώρα η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, η κυρία Καριμάντελη έχει το λόγο, παρακαλώ. Η δημιουργία μιας ε, Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Εργασίας ε, δεν είναι απλά απαραίτητη, είναι αναγκαία. Η κοινωνική Ευρώπη υπάρχει μόνο στα κείμενα, ποτέ στην πραγματικότητα. Φτάνει πλέον. Ας αποκτήσουμε τα μέσα να εφαρμόσουμε το νόμο και να δώσουμε επιτέλους τέλος στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Η αρχή αυτή θα βοηθά όχι μόνο τους αποσπασμένους εργαζομένους αλλά και τους ανθρώπους που εργάζονται σε ένα άλλο κράτος μέλος και κατοικούν εκεί. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πραγματικά να δράσει προς υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να γίνονται σεβαστά η, πραγματική, η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων να αποτελεί πραγματικά ευκαιρία. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα μπορεί να οργανώνει επιθεωρήσεις σε όλη την επικράτεια και να ε, φροντίζει να επιβλέπει την τήρηση όλων των προτύπων σε όλη την Ευρώπη. Ε, έτσι θα εφαρμοστούν ε, τα κοινωνικά δικαιώματα που υπάρχουν μεν επί χάρτου, αλλά δεν τηρούνται στην πραγματικότητα και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ελπίζω, συναδελφοί, να υπερψηφίσουμε με μεγάλη πλειοψηφία το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ένα λεπτό για τον κύριο Τζαμπάσκι για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Για άλλη μια φορά παρατηρούμε ότι η χειραγώγηση καλά κρατεί όσον αφορά ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων και τώρα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αρχή που θα παρεμβαίνει στα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά θα επιβάλλει κυρώσει και στα κράτη-μέλη. Αναφέρονται οι οδικέ μεταφορέ ρητά στην έκθεση, το οποίο σημαίνει ότι οι κυβερνήσει τη Δυτική Ευρώπη εξακολουθούν να φοβούνται του επιχειρηματίε ε, τη Ανατολική Ευρώπη και προσπαθούν να εισάγουν όλο και περισσότερου ε, κανόνε και νόμου. Η αρχή εργασία είναι σημαντική ε, για ολόκληρη την Ένωση. Για να ρυθμιστούν αυτέ οι εργασιακέ σχέσει όμω, πρέπει να διασφαλίζουμε την ελεύθερη επιχειρηματικότητα. Εάν δημιουργηθεί αυτή η αρχή, θα αποτελέσει άλλη μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση να την ε, εγκαταστήσει σε κάποιο κράτος μέλος ε, όπου δεν υπάρχουν άλλες ε, αρχές και η Βουλγαρία είναι μια τέτοια χώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Πάβελ, έχετε το λόγο εκ μέρους της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να χαιρετήσω δύο φίλους που παρακολουθούν τη συζήτηση. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την πρόταση και ευχαριστώ όλους για τις προσπάθειες που έγιναν το τελευταίο έτος. Θα ήθελα να ε, συγχαρώ και την Ρουμανική Προεδρία και τον εισηγητή γιατί καταφέραμε να το κλείσουμε όλο αυτό το θέμα σε λιγότερο από ένα χρόνο. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Εργασίας θα έχει ε, θα χαρακτηρίζεται από μια σημαντική αποστολή και η Κομισιόν ανέφερε ήδη κάποια από τα προβλήματα τα οποία θα λυθούν χάρη στη δημιουργία αυτής της αρχής. Αυτό που θα ήθελα να δω εγώ θα ήταν ε, η αρχή αυτή να εγκατασταθεί στη Ρουμανία. Έχουμε και κάποια επιχειρηματολογία υπέρ αυτού. Έχουμε στη Ρουμανία ένα σύστημα που παρέχει διαφάνεια όπω σε κανένα άλλο κράτο μέλο. Δίνουμε τι ταχύτερε απαντήσει που μπορείτε να φανταστείτε στα αιτήματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία ή τη, ε, τα στοιχεία που αφορούν την απόσπαση των εργαζομένων. Και θεωρούμε ότι αυτό μα ε, καθιστά ικανού. Αποτελεί εγγύηση το ότι αν ε, τα κεντρικά αυτής της αρχής ε, εγκατασταθούν στην Ρωμανία θα έχει μεγάλη επιτυχία στις εργασίες Σας Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σολέ, την Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας ε, θα προωθήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως επίσης και την εφαρμογή των διατάξεων του, του δικαίου της εργασίας για όλους όσοι εργάζονται και έχουν δικαίωμα στην ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Όμως κάποιες από τις προτάσεις της γνωμοδότησής μας έχουν αφαιρεθεί. Παραδείγματος χάρη η εισαγωγή ενός ε, ε, Μια ρήτρα για την ε, συμπερίληψη του, των θεμάτων του, ε, του φύλου, όπως επίσης, η, όπως επίσης και να ληφθούν υπόψη από την Eurostat όταν κάνει στατιστικές εκτιμήσεις, όπως επίσης και θέματα που αφορούν το φύλλο και τέλος να εξασφαλιστεί η ισορροπία των φύλων στη σύνθεση στα όργανα της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Σαφώς ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα επιτύχει και θα αρχίσει να λειτουργεί το ταχύτερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καζά για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον συγητή για το εξαιρετικό αποτέλεσμα του νομοθετήματος αυτό ε, για μια πιο δίκαιη και πιο κοινωνική Ευρώπη. Είναι μια ακόμα επιτυχία κατά την εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Επίσης, είναι επιτυχία λόγω των ευκαιριών που προσφέρει η νέα αγορά. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα βοηθήσει και θα ενισχύσει τις διάφορες αρχές των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν την κατάχρηση και την απάτη και να διευκολύνουν την κινητικότητα προς όφελος των πολιτών. Επίσης, θα ενισχύσει τη συνεργασία ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες και να ενισχύσει την εφαρμογή των νόμων. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργηθούν ξεκάθαροι και δίκαιοι κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται σωστά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την καλή συνεργασία ανάμεσα στις ε, αρχές των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ο σημαντικός ρόλος των κοινωνικών εταίρων στην όλη αυτή διαδικασία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η κοινή αγορά είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και του σχεδίου. Η κινητικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικότητα την οποία διαπιστώνουμε και βιώνουμε καθημερινά. Εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών εργάζονται, ζουν και ταξιδεύουν στις ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ. Εκ μέρου των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ε, κυρία Επίτροπε. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας καλείται να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στο να δώσει ένα τέρμα στην εκμετάλλευση της εργασίας και να εξασφαλίσει σωστή κινητικότητα των εργαζομένων, όπως επίσης και να αντιμετωπίσει το θέμα της ε, αδήλωτης εργασίας. Και αυτό αποτελεί ορόσημο. Η έκκληση που έκανε πέρυσι το Σεπτέμβριο του 2017 συγκεκριμένο πρόεδρος Γιούγκερ, οδήγησε σε μια πρόταση από την Κομισιόν ήδη από το Μάιο πέρυσι για και εντατική εργασία από αυτό το Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο για, τους διάφορους, ε, ε, για τα διάφορα θεσμικά όργανα ε, υπάρχει πεποίθηση ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το σημείο αυτό κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Αρχίζει να σκεφτούμε για λίγο ποιο είναι ο βασικός λόγος συγκεκριμένα ότι όλο και περισσότερο συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει ταχεία και αυξανόμενη ανάγκη επίγουσα και αυξανόμενη ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι βαριές παραβιάσεις μερικών από τα πιο σημαντικά δικαιώματα κάθε Ευρωπαίου πολίτη, τη ελευθερία κίνησης όλη την Ένωση υπό συνθήκες δίκαιη εργασιακή κινητικότητας. Αγαπητοί συνάδελφοι, του τελευταίου μήνε και χρόνια, όλο και περισσότερο μας απασχολεί το θέμα τη ανάπτυξη τη Ένωση ε, υπό το, βάρος των εσωτερικών, οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων. Ε, ε πιστεύω είναι σημαντικό αυτός ο οργανισμός να, δημιουργηθεί το φθινόπωρο και να προβληθεί ως δέσμευση για τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης που θα προσφέρει ζωή με αξιοπρέπεια και ασφάλεια και στην Ένωση θα προσφέρει ε, έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τους δύσκολους καιρούς και θα ήθελα στο τέλος και εγώ να ε, ευχαριστήσω όπως και, ο, όπως και οι άλλοι τον συνάδελφο κύριο Λένερς για το εξαιρετικό ε, έργο του την Επιτροπή και την Επίτροπο, όπως και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχία αυτού του νομοθετήματος. Ευχαριστώ. Η κυρία Άκιν για δύο λεπτά. Χάρκιν για δύο λεπτά, εκ μέρου τη ΑΛΤΕ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την επικοδομητική του προσέγγιση, του σκιώδη ομιλητέ, όπω επίση και την κυρία Τάισον στην Κομισιόν. Θα ήθελα, όταν να πω ότι όταν ε, πρωτοείδα την, την πρόταση είχα κάποια ερωτηματικά σχετικά με την αξία, την προστιθέμενη αξία και ε, ε, τα θέματα της αδειλώτης εργασίας κλπ. Πιστεύω όμως ότι το νομοθέτημα που βρίσκεται τώρα ενώπιόν μας έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία και έχει εξορθολογιστεί ώστε να μας δώσει έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό οργανισμό. Τα άλλα θα επιληθούν διάφορα προβλήματα ε, τα οποία μας απασχολούσαν. Η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων λειτουργεί. Όμως, κατά καιρού προκύπτουν ζητήματα που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη που υπάρχει προς το σύστημα και όπως επίσης τη δικαιοσύνη και τη συμμόρφωση. Αυτά τα θέματα θεωρώ απαιτούν μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα ενισχύσει την λειτουργική συνεργασία και τον συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να διευκολύνει την, ε, την επίλυση των διαφορών. Θεωρώ ότι αυτό το τελικό νομοθέτημα αντιμετωπίζει πολλά από τα προβλήματα που δεν έχουν εντοπιστεί σχετικά με την καθημερινή ε, πράξη Τη ελεύθερη διακίνησης των εργαζομένων. Και με αυτόν τον τρόπο η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων θα υπάρχει για όλους, θα είναι πιο εξορθολογισμένη λόγω της εργασίας μεταξύ των κρατών μελών και κυρίως θα βοηθήσει στην αποκατάσταση τη εμπιστοσύνης προς το σύστημα, την εμπιστοσύνη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ανάμεσα στους πολίτες. Αυτό αυτή δεν θα είναι η τελική μου παρέμβαση του Κοινοβούλου, αλλά είναι μια από τι τελευταίε. Και χαίρομαι ότι σήμερα μπορώ να πω ότι συμμετείχα στην ομάδα η οποία κατάφερε να προχωρήσει ένα νομοθέτημα που θα ενισχύσει την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει προ του πολίτε και τα κράτη-μέλη ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο μπορούν να πιστέψουν και να εμπιστεύονται. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, κυρία Κάρη. Ένα μισή λεπτό τη Ευχαριστώ. Και όσου μίλησαν προηγουμένω και τον εισηγητή, πολλοί κόσμοι αντιμετωπίζει άδικε συνθήκε εργασία, χαμηλέ αμοιβέ, κακέ συνθήκε εργασία, απουσία συμβάσεων, κανένα δικαίωμα. Συχνά πρέπει να δουλεύουν δύο και τρει δουλειέ για να τα βγάλουν πέρα. Το κοινωνικό dumping είναι η σκοτεινή πλευρά τη ενίας αγορά. Η εσωτερική αγορά δίνει προτεραιότητα στα δικαιώματα των επιχειρήσεων και στα κέρδη αντί να δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους. Η ενιαία αγορά απομακρύνει τις αγορές από τους ανθρώπους, από ε, τους τοπικούς πολιτικούς, από τη δημοκρατική λογοδοσία. Χιλιάδες άνθρωποι ζουν καθημερινά τις συνέπειες όλων αυτών και απαιτούν λύσεις. Από εμάς απαιτούν να κάνουμε κάτι αποτελεσματικό κατά του κοινωνικού ντάμπινγκ ώστε να διασφαλίζονται αυτές οι συνθήκες εργασίας ε, και τι απάντηση τους δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αντλεί πόρους ε, για να υποστηρίζει τη γραφειοκρατία της. Ε, ενώ η σωστή απάντηση θα ήταν λιγότερη Ευρωπαϊκή Ένωση και περισσότερη εξουσία στους πολίτες. Αλλά εμεί ε, ενδυναμώνουμε διαρκώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι λάθο απάντηση. Δεν χρειάζονται περισσότερε αρχέ και οργανισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, χρειάζονται τι ε, αγορέ λίγο να, να ε, κάνουν άκρη για να προστατευθούν τα δικαιώματά του. Η κυρία Άουκεν, εκ μέρου των Πρασίνων. Χαίρομαι ιδιαίτερα που τώρα έχουμε περισσότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αρχή για την αγορά εργασίας που θα μπορέσει να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να δώσουν τέλος σε ζητήματα όπως το κοινωνικό ντάμπινγκ μέσω για παράδειγμα επιθεωρήσεων. Εκατομμύρια Ευρωπαίοι εργάζονται σε χώρες ε, διαφορετικές από τη δική του συμβάλλουν ε, στην κοινωνική προστασία και στην κοινωνική ασφάλιση και στο, ε, με τους φόρους τους αλλά δεν εργάζονται υπό σωστές συνθήκες ο κόσμος εργάζεται για να τα βγάλει πέρα όχι για να κλέψει είναι σημαντικό λοιπόν να ασχοληθούμε με τις διασυνοριακές για παράδειγμα περιπτώσεις ε, Έχουμε την υπόθεση των 200 οδηγών από τι Φιλιππίνες που ζουν και εργάζονται υπό συνθήκες Σκλαβιά. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνθήκε και προστασία ε, χρησιμοποιώντας το, δανικό, το δανέζικο σύστημα ε, πρόνοιας ως πρότυπο ε, και να δώσουμε και το δικαίωμα στους Ευρωπαίους πολίτες να μπορούν να καταγγέλουν απευθείας τις καταχρήσεις είναι πολλά στοιχεία αυτής της πρότασης τα οποία θα έχουν την υποστήριξή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Παπαδάκης για ένα λεπτό παρακαλώ. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στην Ελλάδα για να ελέγξει όλους τους χώρους δουλειάς μια φορά τουλάχιστον χρειάζεται 13 ολόκληρα χρόνια ευρωπαϊκή ένωση και κυβερνήσεις ρήμαξαν και αυτούς τους ελάχιστους και ανεπαρκείς κρατικούς ελεκτικούς μηχανισμούς. στόχος αποτελεί η εργοδοσία με λιμένα χέρια να ξεζουμίζει ανεμπόδιστα τους εργαζόμενους. σε αυτά τα συντρίμμια των επιθεωρήσεων εργασίας σε κάθε χώρα έρχεται να συγκροτηθεί η λεγόμενη ευρωπαϊκή αρχή εργασίας. στόχος του νέου ευρωμηχανισμού είναι να πολλαπλασιάσει την κινητικότητα των εργαζομένων γιατί όπω προκλητικά η ευρωπαϊκή ένωση αναφέρει μόνο 700.000 εργαζόμενοι μετακινούνται ετησίω από χώρα σε χώρα. προστατεύεται δηλαδή και προωθείται την εργασιακή γαλέρα τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία με βάση τον αντεργατικό ευρωπαϊκό πυλώνα τον οποίο συνυπέγραψαν σύριζα νέα δημοκρατία και κοινάλ στην ελλάδα προωθείται η αντικατάσταση των συλλογικών συμβάσεων με εργατικά δικαιώματα ακόμα πιο κάτω στον αδύρ που βαφτίζονται ελάχιστοι κανόνε. κριτήριο ψήφου και αυτά για τους εργαζόμενους με την ταξική οργάνωση και ισχυρό ΚΚΕ παντού να αντεπιτεθούν να βάλουν εμπόδια στην εργασιακή ζούγκλα της ευρωπαϊκής ένωσης. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. Η κινητικότητα είναι θεμελιώδες δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε αποσπασμένους εργαζόμενους, μεθοριακούς εργαζόμενους και διάφορους ανθρώπους που μπορεί χρόνια ολόκληρα να δουλεύουν σε διαφορετική χώρα από την πατρίδα τους. Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν συζητήσει επανειλημμένα και επιμακρών τα θέματα της κινητικότητας των εργαζομένων, δέσμες μέτρων κινητικότητας, οδηγία για την απόσπαση, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης κτλ. Μα ενδιαφέρει λοιπόν η συνεργασία των κρατών μελών ε, για την καταπολέμηση της αδήλωτη εργασίας και των αθέμητων πρακτικών. Πολλές φορές συζητήσει ήταν και πολύ έντονες και πολύ ε, Υπάρχουν πολλά προβλήματα γιατί είναι πολύ περίπλοκη η νομοθεσία αυτή τη στιγμή. Η ιδέα λοιπόν ίδρυση, μια Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ε, ε, που θα βοηθήσει τους εργαζομένους να καταλάβουν τι δικαιώματα έχουν και τι υποχρεώσεις είναι σημαντικό και χρειαζόμαστε μια τέτοια αρχή εργασίας. Κάποιοι είπαν να έχει ισχυρές ελεγκτικές εξουσίες η ε, αρχή εργασίας. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Είμαι πάρα πολύ υπέρ της ε, υποστηρικτικής λογικής, αλλά πολύ αντίθετη με την ελεγκτική αρχή. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι και οι εταιρείε να μάθουν τι δικαιώματα έχουν και πώς θα τα εφαρμόζουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρέσο, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ. Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της ομάδας μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πρώτο αποτέλεσμα της έγκρισης του πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Εδώ και χρόνια κάνουμε αγώνε προ αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δείχνει ότι ο στόχο μα για την κοινωνική Ευρώπη είναι σωστό. Δεν περιορίζεται στα προγράμματα, αλλά παρεμβαίνει πραγματικά για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών και να του βοηθήσει στην αναζήτηση εργασία. Η νέα αρχή θα αποτελήσει σημαντικό εργαλείο. Θα διασφαλίσει τη μέγιστη προστασία, αξιοπρέπεια, ισοτιμία ε, στου εργαζόμενου που κινούνται εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και στου διασυνοριακού εργαζομένου. Θα υποστηρίσει τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση του κοινωνικού ντάμπινγκ, της μαύρης εργασίας ε, και θα παράσχει συνοχή στους ε, θέματα τη αποσπάσης εργαζομένων. Υπενθυμίζω στην Κομισιόν ότι το Κοινοβούλιο, για το Κοινοβούλιο θα είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε στην επιλογή της έδρας, διότι όπως και για την αίμα είμαστε συναρμόδιοι για τη χρηματοδότηση, οπότε είμαστε συναρμόδιοι και για την επιλογή εγκατάσταση. Ευχαριστώ κυρία Μπρέσο. Ο κύριος Καλβετσόμπο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρία Επίτροπε, για άλλη μια φορά θα μιλήσω εγώ. Τι να κάνουμε Είμαι εθισμένος στις κοινωνικές πολιτικές και στην ε, κοινωνική Ευρώπη. Θέλω να πω μόνο ότι αυτό εγγράφεται στη γραμμή των όσων είπε ο Επίτροπος ε, καταλήγοντας την προηγούμενη συζήτηση. Καταβάλουμε μια μεγάλη προσπάθεια τώρα στο τέλος της θητείας. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο και λίγο πιο διστακτικά το Συμβούλιο πορευόμαστε προς τη δημιουργία της κοινωνικής Ευρώπης και τη θετική της εξέλιξη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και όλους τους σκιώδεις για το έργο τους. Προφανώς θα μπορούσε να είναι τέλειο, που δεν είναι, αλλά είναι ένα τεράστιο βήμα προς τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, προς την επαγρύπνηση για να εντοπίζονται οι καταχρήσεις και να εφαρμόζονται τα ελάχιστα δικαιώματα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε παρά να καλωσορίσουμε ένα τέτοιο εγχείρημα από το Κοινοβούλιο και να το υποστηρίξουμε. Ο κύριος Βάνταν Κέντελαρ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο θέμητος ανταγωνισμός στην αγορά εργασίας μεταξύ ε, ημεδαπών και αλλοδεπών συναδέλφων είναι κάτι που ο κόσμος ε, μου αναφέρει συχνά η διασυνοριακή απάτη στα κοινωνικά ζητήματα φτάνει κάθε μέρα στους πολίτες μας. Ξέρουμε όμως τι πρέπει να κάνουμε. Είναι πολύ σαφή τα ελλείμματα. Το πρόβλημα είναι στα κράτη-μέλη που είναι απρόθυμα ε, να κάνουν κάτι για τον ουσιαστικό έλεγχο. Και ποιο είναι το ικτρό αποτέλεσμα. Σιγά σιγά χάνεται η εσωτερική αγορά και η υποστήριξή της ενώ ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ. Στη δική μου περιφέρεια, στη Δυτική Φλάνδρα, εναγωνίω ζητούν οι εταιρείε εργαζομένου και του υποδέχονται με ανοιχτέ τι αγκάλε. Η ε, κινητικότητα τη εργασία υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία. Αλλά για να είναι βιώσιμη, ε, θα πρέπει να γίνεται με τρόπο σωστό και συντεταγμένο και δίκαιο. Και εκεί χωλαίνει η υπόθεση. Πολλοί ε, πολίτε θεωρούν ότι υπάρχουν διάφοροι καουμπόιδε που έρχονται και αλωνίζουν ατιμωρητοί δεν τιμωρούνται ε, οι παραβάτες. Ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας λοιπόν πρέπει να έρθει να φέρει αλλαγές γρήγορα ε, και αποτελεσματικά να πληροφορούνται οι ενδιαφερόμενοι. Συνάδελφοι, στην αρχή της θητείας αυτής ε, μας υποσχέθηκαν τριπλό α στη κοινωνική βαθμολογία. το ένα α τώρα είναι Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και χάρη στην κυρία Τέισεν θα πρέπει να βοηθήσουμε τους πολίτες να ξεφύγουν από την απογοήτευση και να πιστέψουν και πάλι στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαλάς, για ένα λεπτό παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Επίτροπε. Ναι, πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Πρόκειται για ένα βήμα προς τα εμπρός. Σημαντικό Ωστόσο, όπω γνωρίζουμε, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε διαδικασία συνδιαλλαγή όσον αφορά το σύστημα τη ρύθμιση, για παράδειγμα, και τη καταπολέμηση τη απάτη. Γι' αυτό το λόγο θα χρειαστούν και άλλα βήματα προ τα εμπρό. Και κατά την άποψή μου, είναι τρία αυτά τα βήματα. Πραγματική ευρωπαϊκή επιθεώρηση τη εργασία που θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσει ε, στου παραβάτε, όχι μόνο οικονομικέ, όπω ήδη συμβαίνει ενίοτε σε εθνικό επίπεδο, αλλά και ποινικέ διότι ξέρουμε ότι από αυτή την άποψη ο φόβο πρέπει να αλλάξει στρατόπεδο και ορισμένοι παραβάτε σήμερα που οργανώνουν το κοινωνικό dumping θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πράττοντας αυτό θα καταβάλουν προσωπικά το τίμημα. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να θέσει επί χάρτου μια ηλεκτρονική κάρτα κοινωνική ασφάλισης που θα αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο φορητότητα των δικαιωμάτων. Ένα πρώτο βήμα λοιπόν ε, και άλλα βήματα θα ακολουθήσουν ώστε το κοινωνικό ντάμπινγκ να αποτελεί μια πια κακή ανάμνηση και όχι πραγματικότητα. Κυρία Ιλφσκοκ, για ένα λεπτό. Thank you. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δουλέψει πολύ για την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων και υπήρξε μεγάλη επιτυχία για πολλούς ε, εργαζομένους και για τα συνδικάτα. Ε, ναι, πράγματα χρειάζεται ίση αμοιβή για ίση εργασία. Τώρα πρέπει να υλοποιήσουμε επιτέλους αυτή την οδηγία και σωστά μάλιστα στα κράτη-μέλη. Πρέπει να υπάρχει και παρακολούθηση. Αυτή η αρχή λοιπόν, η εν λόγω αρχή, είναι ένα καλό φορέα που θα παρακολουθεί την εφαρμογή τη αποσπάση των εργαζομένων. Πρέπει να υπάρχει σωστή ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μέλων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλέ παραβάσει σε θέματα κοινωνική ασφάλιση. Χωρί ενημέρωση είναι αδύνατο να διορθωθεί η κατάσταση, χωρί να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Οι εργαζόμενοι στην Ευρώπη πρέπει να είναι διασφαλισμένοι. Πρέπει να εξασφαλίζουμε στους πολίτες ε, ότι υπάρχει ασφάλεια. Ε, δεν ε, πρέπει να ζουν χειρότερες συνθήκες όταν μετακινούνται σε άλλη χώρα. Και χαίρομαι που έχουμε ένα συμβιβασμό που ε, υποστηρίζει τα εθνικά προνόμια μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία. Κατά τη διάρκεια αυτή τη θητεία ήταν πολύ σημαντική. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πέντε συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο στη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΙ. Βλέπετε να καταφθάνουν οι συνάδελφοι, άρα γίνεται λίγη φασαρία. Παρακαλώ να μιλάτε λίγο δυνατά όσοι πάρετε το λόγο. κυρία Σόιντροβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Επίτροπο και να της ευχηθώ καλή επιτυχία, καθώς επίσης και τον εισηγητή μας, τον κύριο Λέναρς. Είναι καλή η συμφωνία που επιτεύχθη τελικώς. Ε, γενικά δεν είμαι υπέρ της δημιουργίας νέων ευρωπαϊκών οργανισμών, αλλά η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Αρχή έχει πραγματικά τη δυνατότητα να λύσει σε κάποιο βαθμό τις διαφορές και τις δυσκολίες που έχουμε στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ε, σε τομείς που ακόμα αυτό δεν έχει γίνει δυνατό. Ας πούμε, ε, καταπολέμηση των καρτέλ. Δεν εφαρμόζονται σωστά όλες οδηγίες σε όλα τα κράτη-μέλη για την καταπολέμηση ε, και το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος κτλ. Δεν θα πρέπει λοιπόν όμως να έχουμε επικαλύψεις τώρα με το έργο άλλων οργανισμών και αρχών. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι επιθεωρητές ε, θα συμμετέχουν εκεί εθελοντικά και τα κράτη-μέλη θα σέβονται την ε, ανεξαρτησία της αρχής. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ, έχουμε και άλλους συναδέλφους που θα πάρουν το λόγο ησυχία όσο γίνεται. Η κυρία Τόμασιτς. Μικρόφωνο. Αν μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο, εντάξει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στηρίζω τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη δημιουργία ενός κλίματος εργασίας όπου θα είναι φυσιολογική τήρηση αυτών των δικαιωμάτων. Σε κάποιες περιφέρειες της Ευρώπης αυτό δεν ισχύει παρά την καλή νομοθεσία και την γραφειοκρατία η οποία τους ενισχύει. Πώς είναι αυτό δυνατόν. Υπάρχουν διοικητικέ αρχές που δεν αποτελούν εγγύηση για την τήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά αντίθετα όσο περισσότερη νομοθεσία και γραφειοκρατία υπάρχει, τόσο πιο περιορισμένη είναι η προστασία των εργαζομένων. Δεν στηρίζω αυτή την αρχή, διότι συνεπάγεται περισσότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ε, καταπολέμηση ε, κατά των μη αποτελεσματικών εθνικών οργανισμών. Κάποιος θα πρέπει να το πληρώσει αυτό, θα, θα είναι εργαζόμενοι, δεν θα ωφεληθούν καθόλου από αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Κούνεβα, παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάντε λίγη ησυχία σας, παρακαλώ. Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας αυτός ο τίτλος ακούγεται πολύ ωραία αλλά τι λέμε εδώ σε χιλιάδες εργαζομένους που δουλεύουν απλήρωτοι χωρίς κοινωνική ασφάλεια συχνά και χωρίς ασφάλιση επαγγελματικού κινδύνου. οι πολίτες μας πέφτουν κατά χιλιάδες θύματα των σύγχρονων δουλεμπορίων στην ευρωπαϊκή ένωση και δεν χρειάζεται τα καλά λόγια μας. τα σωστά μέτρα χρειάζονται πότε θα έχει αξία μια νέα αρχή εργασίας όταν δεν θα κάνει μόνο έλεγχο και καταγραφή των παραβιάσεων αλλά θα προφυλάσσει πραγματικά τους εργαζόμενους από τους εργοδότες που ψάχνουν τα τίματά τους στη διασυνορική απασχόληση δηλαδή μια ευρωπαϊκή αρχή για την εργασία που παρίσταται και στα δικαστήρια στο πλευρό των εργαζομένων ώστε να γίνει το ευρωπαϊκό στήριγμά του. ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γιασλοβέσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό, η αρχή... Ε, ησυχία παρακαλώ λέει η πρόεδρος. Λοιπόν, η επίτροπο τόνισε ε, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ε, για τους ε, ανθρώπους που προσλαμβάνουν ανθρώπους εντός της ενίας αγοράς, τη συνεργασία μεταξύ αρχών των κρατών μελών, αλλά αυτό δεν είναι παρά ένα μέρος των αρμοδιοτήτων της νέας αρχής, η οποία θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα προστατευτισμού και λάθος παρανοήσεις της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη. Η αποτελεσματικότητα θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα του Διευθυντή και του Συμβουλίου και